και την έκθεσή του που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέρημνας για την, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών. Για να ξεκινήσουμε έχει το λόγο ο κύριος Τοντέους Τσβίφκα, εισηγητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι παρόλο που ασχοληθήκαμε με την αναδιατύπωση αυτού του συγκεκριμένου κανονισμού, ε, συνεχίζουμε να επεξεργόμαστε το ειδικό νομοθετικό καθεστώς ε, που ε, αφήνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε απλό συμβουλευτικό ρόλο, στην απλή διαδικασία διαβούλευσης, ενώ το Συμβούλιο με την ανάγκη ομοφωνίας παραμένει ο μοναδικός νομοθέτης στην περίπτωση αυτή ενώ εμείς με μεγάλο ενθουσιασμό ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό και νομίζω ότι πραγματικά κάναμε πολύ καλή δουλειά. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από τις ευχαριστίες. Ευχαριστίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση, πολύ καλή πρόταση αναδιατύπωσης για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ιδιαίτερα τους όδης συζητητές με τους οποίους είχα αγαστή συνεργασία που με γέμισε με ικανοποίηση. Ήταν πολύ άρτια η συνεργασία μας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν μεν καλή, αλλά παρόλα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε και τις δικές του τροπολογίες που πιστεύω ακράδαντα ότι πραγματικά βελτιώνουν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα προ παροτρύνουν το Συμβούλιο να λάβει υπόψη και τα δικά μας σχόλια. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν το θέμα της ακρόασης του παιδιού. Για μας ε, το ζήτημα αυτό έχει κέρια σημασία στον ε, κανονισμό, γιατί θεωρώ ότι σε επίπεδο διαφοράς αγωνικής μέρημνα για θέματα επιμέλεια ε, ή σε περίπτωση απαγωγή του παιδιού, Δυστυχώ, το παιδί είναι το πιο αδύναμο και βάλω το μέρος της ε, όλης αντιδικίας και θα πρέπει να το προσέξουμε, να το προστατεύσουμε, ε, να λάβουμε υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του και θα πρέπει να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ε, θέση του παιδιού σε αυτή την αντιδικία. Φυσικά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την ακρόαση του παιδιού σε κάθε περίπτωση. Αυτό εξαρτάται από το δικαστή. Αυτός έχει τη διακριτική ευχαίρεια. Αυτό που προσθέτουμε ως καινοτομία είναι η ανάγκη αιτιολόγησης σε περίπτωση απόρριψης της ακρόασης του παιδιού. Επίσης, ε, τονίζουμε ότι τέτοιου είδους ακροάσεις θα πρέπει να τηρούν κάποιες κοινέ προδιαγραφές και πρότυπα, να δημιουργηθεί μια φιλική, μια πρόσφορη ευνοϊκή ατμόσφαιρα για το παιδί, ένα καλό κλίμα. Επίσης θα πρέπει η ακρόαση να γίνεται από έναν ειδικά καταρτισμένο δικαστή ή εμπειρογνώμονα χωρίς την πίεση, την παρουσία τρίτων ή χωρίς πίεση η συμμετοχή των ε, γονιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να γίνεται ανεπηρέαστα για το παιδί ακρόαση. Επίσης, η άσκηση της γονικής μέρημνας είναι σημαντικό θέμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα της χρήσης της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου διευθέτησης ε, διαφοράς γιατί με τη διαμεσολάβηση θα έχουμε σύντμηση της διαδικασίας, μια πιο ήπια, μια πιο ήπια διαδικασία και επίσης μια λιγότερο δαπανηρή διαδικασία. Ε, και σε περίπτωση που ο δικαστής αποφασίσει την ανάθεση του παιδιού σε θετή οικογένεια ή σε κάποιο ίδρυμα ή σε κάποιο κέντρο, κατέθεσα τη δική μου πρόταση που υποστήριξε και η νομική επιτροπή. Θα πρέπει να λάβει ο δικαστής ο αρμόδιος φορέας τη δυνατότητα να παραμείνει το παιδί ε, στη χώρα που εκδικάζεται η απόφαση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σε περίπτωση που είναι χρονοβόρε οι διαδικασίε. Επίση, χαιρόμαστε για την κατάργηση τη ε, διαδικασία κήρυξη τη εκτελεστότητα του εξεκουάτορ. Δεν χρειάζεται πια τέτοια διαδικασία ε, κήρυξη εκτελεστότητα για αποφάσει που έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη-μέλη. Και σα ευχαριστώ που επιτρέψατε την ε, σημείωση κάποιο πρόοδου για το θέμα αυτό. Θα παρακολουθήσω με προσοχή τη συζήτηση και θα δευτερολογήσω στο τέλο. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Αβραμόπουλο τώρα έχει το λόγο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <clears throat> Uh, honorable members of the Parliament, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η ανακοίνωση Βρυξέλλες 2α είναι ε, ο οδηγός ε, για θέματα γαμικών ε, διαφορών. Είναι ο οδηγός εκείνος που προσφέρει την προστασία στα παιδιά. Η αναθεώρηση αυτού του κανονισμού αντιμετωπίζει τις ε, αδυναμίες που υπάρχουν σχετικά με την γονική μέρημνα. Αυτά κατά το παρελθόν επισημάνθηκαν από τους αξιότιμους βουλευτές. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν ένα κοινό στόχο. Επιθυμούμε να εμποδίσουμε έτσι ώστε σε ε, περιπτώσεις ε, διασυνοριακών διαφορών τα παιδιά να καθίσανται όμοιροι μακροχρόνιων διενέξεων. Επίσης θέλουμε να διευκολύνουμε τις ε, διαδικασίες για τις οικογένειες με διάφορους τρόπους. Μεταξύ άλλων περιορίζοντας ε, την διάρκεια και το κόστος αυτών των διαδικασιών. Πριν λοιπόν αναφερθώ στις τροπολογίες σας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας ε, στον εισηγητή, τον κύριο Ζήφκα, για την ε, εξαιρετική συνεργασία που είχαμε σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που η έκθεση αναγνωρίζει το ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να επιστρέφουν ομαλά τα παιδιά στις οικογένειες. Αυτό είναι προς το συμφέρον των παιδιών και προς το συμφέρον της σχέσης με τους γονείς. Ε, ιδιαίτερα χαιρετίζω τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση που αποσκοπούν στο να περιορίσουν ε, ουσιαστικά την ε, τις αρνητικές επιπτώσεις ε, στα παιδιά τα οποία πήχτησαν από έναν γονέα, από έναν από τους γονείς. Αυτά συμβαδίζουν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέτρα αυτά στην πράξη θα περιλαμβάνουν λιγότερο επίπονες διαδικασίες για τους γονείς ταχύτερη λήψη αποφάσεων από τους δικαστές σε περιπτώσεις ε, διασυνοριακές. Ε, και θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θα ανακτήσουν την σταθερότητα που χρειάζονται, θα μπορούν να επιστρέψουν γρηγορότερα στην ε, οικογενειακή ζωή η διευκόλυνση της εφαρμογής των αποφάσεων των δικαστών αυτό είναι ένα άλλο καθοριστικό στοιχείο για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των παιδιών και των οικογενειών τους. Η κατάργηση τις ε, διαδικασίες ε, διαμεσολάβησης για να εφαρμόζονται οι διασυνοριακές ε, αποφάσεις, για να εφαρμόζονται διασυνοριακά οι αποφάσεις των δικαστών. Αυτό θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν και οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των αμυνόμενων. Ε, χαιρετίζω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα αυτά τα μέτρα. Όσον αφορά τώρα στις ε, τροπολογίες για τα δικαιώματα των παιδιών, το να εισακούνται τα παιδιά ε, στη διάρκεια της διαδικασίας, ε, λαμβάνω υπόψη μου την επιθυμία του Κοινοβουλίου που είναι να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά να προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι η αναφορά σε πρακτικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ακρόαση. Εμείς αξιολογήσαμε αυτή τη δυνατότητα. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι υπάρχοντες κανόνες και οι πρακτικές στα κράτη-μέλη ε, σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα αποκλίνουσες, θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματικότερο να ε, εφαρμόζουμε υπάρχοντες κανόνες που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών, μια σύμβαση ε, την οποία έχουν ήδη υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν αυτός ο ιδιαίτερος κανόνας να γίνει αποδεκτός ε, κυρίως στην τελευταία του εκδοχή. Όπως όλοι σας γνωρίζετε, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρότασή μας στον τομέα αυτό θα διασφαλίσει τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να ακούει την άποψή τους ε, στι ε, διαδικασίε, δικαστικές διαδικασίε. Η αμοιβαία αναγνώριση των πρακτικών των κρατών μελών επ' αυτού του θέματος θα ε, οδηγήσει στο να αποφεύγονται απορρίψεις και με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να έχουμε την ε, ουσιαστική εφαρμογή αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος της ε, αποτελεσματικότητας και για να αποφεύγονται επικαλύψεις δεν έχουμε συμπεριλάβει ιδιαίτερους κανόνες που να αφορούν ε, στη διαμεσολάβηση για διενέξεις ανάμεσα στους γονείς όπως ακριβώς το ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η υπάρχουσα οδηγία για τη διαμεσολάβηση ήδη καλύπτει αποτελεσματικούς κανόνες και προβλέπει την υποστήριξη προς τους γονείς κατά την επίλυση των διαφορών τους. Τέλος, ε, διαπίστωσα ότι οι τροπολογίες σας εστιάζουν σε στενή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, και εδώ, για άλλη μια φορά, μιλάμε με μία και μόνο φωνή. Οι κεντρικές αρχές ε, είναι η άμεση επαφή των γονέων και γι' αυτό πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή των αποφάσεων των δικαστών. Η έκθεση και οι προτινόμενες τροπολογίες αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για πιο αποτελεσματική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντάλι, εκ μέρου των Αναφορών, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ και τον συγκητή μας. Ε, σήμερα συζητούμε ένα πολύ λεπτό θέμα με ε, άμεση συνέπειες στη ζωή χιλιάδων πολιτών και κυρίως παιδιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι έχουμε καθήκον ε, να εξασφαλίσουμε μια καλόπιστη προστασία, μια, την προστασία για τα παιδιά και όποιους γονείς ε, δρούν καλόπιστα. Υπάρχει περίπτωση απαγωγής από τον έναν εκ των δύο γονέων της βαρός παιδιών και δεν είναι δυνατόν να μείνουμε αδρανείς, γιατί αυτό παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε παιδιού, οπουδήποτε και αν αυτό βρίσκεται. Και όντως αλλάζει ο κόσμος στον οποίο ζούμε και τα θέματα τα οικογενειακά, του οικογενειακού δικαίου ε, αλλάζουν γιατί στο παρελθόν βέβαια αποκλειστικά στο εθνικό δίκαιο ρυθμίζονταν το, ε, οι οικογενειακές διαφορές ενώ τώρα χρειάζεται διεθνής διευθέτηση καθώς είναι και διεθνής και η γάμη αλλά και οι ε, γαμικές διαφορές και οι διαφορές για την επιμέλεια των τέκνων διεθνής. Το δικαίωμα λοιπόν ε, της επιμέλειας ε, πρέπει να, αντιμετωπιστεί κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί ένας γονιός να αφαιρεί το παιδί με απαγωγή από τον άλλο γονιό. Πρέπει να κλείσουμε κάθε παραθυράκι και να φροντίσουμε ο κανονισμός να μην μπορεί να οδηγήσει σε ερμηνείες που να ευνοούν τον γονιό που έχει υπετιότητα για την απαγωγή του παιδιού. Ε, και πρέπει βεβαίως το δικαστηρίο της καταγωγής του παιδιού να είναι εκείνο που θα λαμβάνει τις αποφάσεις, να αποφύγουμε το forum shopping, την επιλογή της ευνοϊκότερης νομοθεσίας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε οποιαδήποτε ε, ζημία ή τραυματική εμπειρία για το παιδί. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και να είναι αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα παρακαλώ τον κύριο Πάβελ Σβόμποντα να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και ιδιαίτερος βέβαια τον εισηγητή μας κύριο Σβέφκα για την δουλειά αυτή στην έκθεση και θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλου του ε, πολίτε ότι όταν κατατίθενται προτάσει, προτάσει μάλιστα νομοθετικέ οι οποίε αφορούν πολλού πολίτε, θα ε, γίνεται η δουλειά με πρώτο μέλημα τα συμφέρον του. 16 εκατομμύρια μεικτέ οικογένειε έχουμε στην Ευρώπη, 140.000 διαζύγια δυστυχώς κάθε χρόνο με διεθνεί διαστάσει και 180.000 παιδιά, 180 ε, παιδιά μάλλον το χρόνο απάγονται από τον, γονέα, από τον Έτσι λοιπόν η εκτέλεση ε, αποφάσεων, ε, είτε πρόκειται για γαμικές διαφορές, είτε πρόκειται για επιμέλεια παιδιών, έχει μεν εγκριθεί ως νομοθέτημα από το 2005 και ισχύει σε όλες τις χώρες πριν της Δανίας, αλλά δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται όλα τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού. Με τον νέο κανονισμό επιδιώκεται η βελτίωση των διατάξεων, των δικονομικών και ε, εγκαθιδρύεται ο σεβασμός στην επικουρικότητα όπως επίσης και ε, η εφαρμογή του κανονισμού αφορά μόνο διασυνοριακές υποθέσεις, δηλαδή υποθέσεις όπου οι γονείς έχουν διαφορετική ηθαγένεια. Μέλημα της Επιτροπής μας και όλου του Κοινοβουλίου είναι να εγκριθεί το νομοθέτημα κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζει τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού. Εξ ονόματος της Επιτροπής ε, των Νομικών Υποθέσεων λοιπόν σας διαβεβαιώ ότι με το κανονισμό αυτό έχουμε δώσει ιδιαίτερο μέλημα για την πτυχή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει η Πρόεδρος και παρακαλώ την κυρία Εύριν Γκέπχαρτ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Σβόμποντα το είπε ήδη ότι σήμερα ε, πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι κατά το παρελθόν ε, χαίρονται και εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως υπάρχουν και ε, μειονεκτήματα γιατί σε τελική ανάλυση δεν στέφονται με επιτυχία όλοι αυτοί οι μεικτοί γάμοι. Εγώ όταν ήμουν διαμεσολαβήτρια βίωσα καταστάσεις όπου παιδιά εμπλέκονται σε τέτοιου είδους προβλήματα και πρέπει να σας πω ότι αυτές είναι πολύ δυσάρεστες ιστορίες αυτό λοιπόν όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και εξεπλάγει πολύ θετικά όταν διαπίστωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα σημαντικό αριθμό των προτάσεων που είχα καταθέσει εγώ για να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα. Τα συμπεριέλαβε στο σχέδιό της και αυτό είναι πολύ θετικό. Ιδιαίτερα λοιπόν το ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία των δικαστηρίων και των αρμοδίων αρχών. Ταχύτερη συνεργασία. Γιατί όσο σέρνονται αυτές οι διαδικασίες, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα, κυρίως για τα παιδιά. Ένας άλλος τομέας, εδώ τρέψτε μου να πω ότι τίθεται και θέμα νομικής ασφάλειας. Άλλος τομέας, ιδιαίτερα σημαντικός, είναι η, το να εισακούται η άποψη των παιδιών. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά από τη Συνθήκη των Εθνών να λαμβάνονται υπόψη, να ακούγεται η άποψη των παιδιών με τα δικά του τα λόγια και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ε, βρίσκονται τα παιδιά σε προστατευμένο περιβάλλον. Εκεί να τους τίθενται ερωτήσει και όχι σε μια αίθουσα που μπορεί να είναι τρομακτική για παιδιά, ας πούμε όχι σε αίθουσα δικαστηρίου. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε να είναι σωστές και οι συνθήκες ε, πλαίσιο, ε, να είναι ικανοποιητικέ οι συνθήκες αυτές για τα παιδιά. Και κάτι άλλο, και εδώ ευχαριστώ θερμά τον κύριο Φσχέσκα γιατί συνεργαστήκαμε πολύ καλά, είναι το θέμα της ε, διαμεσολάβησης. Πράγματι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανόνες για τη διαμεσολάβηση, όμως αυτοί δεν αρκούν, δεν αρκούν βλέποντας ότι τα δικαστήρια δεν εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε για ε, γονείς με περιορισμένους οικονομικούς πόρους ε, οι γονείς αυτοί να μην μένουν μόνοι τους γιατί τα ερωτήματα που τίθενται, τα θέματα της ε, διαμεσολάβησης είναι θέματα που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά κύριε Τσβεύσκα μπορούν να εξοικονομήσουν κόστος. Οι διαδικασίες να είναι ταχύτερες, ίσως να είναι και περιττές οι διαδικασίες και οι διαδικασίες να διεξάγονται με καλύτερο τρόπο και για τους γονείς και για τα παιδιά. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και το τελευταίο που πρέπει να δείξω. Εκεί δυστυχώς διαφωνήσαμε. Ο κύριος Γεύκα και εγώ ε, διαφωνήσαμε και μέχρι τώρα υπάρχει διάσταση απόψεων και στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τα σύμφωνα συμβίωσης και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά ατόμων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και τα παιδιά εντός γάμου. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό γιατί είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Γκέρκ έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν δύο τσακώνονται χαίρεται ο τρίτος. Αυτό είναι μια σοφία, έχει προκύψει από τη ζωή και αφορά τους γονείς που παίρνουν διαζύγιο. Σε μια τέτοια διαδικασία όμως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε κατά νου το καλό του παιδιού. Η Γερμανία σε αυτό το θέμα υπολείπεται. Η δική μας η κυβέρνηση πρέπει να επεξεργαστεί το δίκαιο περί διαζυγίων. Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο όπως και πολλά κράτη-μέλη. Οι πολλές αναφορές που κατατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δουλειά των κοινωνικών λειτουργών μου καταδεικνύει ότι πράγματι χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις. Για πάνω από ένα χρόνο εγώ παρακολούθησα μία Γαλλίδα μητέρα και την κόρη της. Ε, σήμερα βγήκε η απόφαση προ όφελο της, υπέρ της. Γι' αυτό και λέω, η Γερμανία κουνήσου. Ε, εάν κουνηθεί, θα είναι αυτό προ όφελο ε, πολλών οικογενειών. Θα είναι προ όφελο πατεράντων και παιδιών. Η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει πολλά κίνητρα για να κινητοποιηθεί η γερμανική πολιτική. Ας το κάνουμε λοιπόν για το καλό και το συμφέροντα των παιδιών. Η αύξηση του αριθμού των ζευγαριών διαφορετικών εθνικοτήτων καθιστά αναγκαία τη βελτίωση και αποσαφήνιση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή δικαιοδοσία, για την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέρημνας και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην ανασφάλεια δικαίου καθώς και σε περιττές καθυστερήσεις σχετικών υποθέσεων που επηρεάζουν αρνητικά τις εμπλεκόμενες οικογένειες. πρέπει να δίδεται έμφαση στην προστασία του συμφέροντος των παιδιών συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων. είναι επίσης αναγκαία η εξειδικευμένη κατάρτιση των δικαστών και η ενίσχυση του επικουρικού θεσμού της διαμεσολάβησης. χρειαζόμαστε ακόμη συγκέντρωση της δικαιοδοσίας για τις διεθνείς απαγωγές παιδιών σε εξειδικευμένα δικαστήρια και εξορθολογισμό των λόγων τυχόν άρνησης εκτέλεσης σχετικών αλλοδαπών αποφάσεων. με βάση τις παραμέτρους αυτές συμφωνώ με την έκθεση του ευρωβουλευτή κ. τσβίφκα που συζητούμε σήμερα και θα την υπερψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φεράρα από την ε, ομάδα EFDD. Η πρόταση για αναδιατύπωση του κανονισμού έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. βεβαίω, η αναγνώριση, η διευκόλυνση αναγνώριση ε, των αποφάσεων και τη αντιμετώπιση των προβλημάτων ε, σε σχέση με τους ανήλικου. με ε, κύριο γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου πρέπει να επικρατούν σε σχέση με άλλα δικαιώματα. Σημασία έχει και η ειδική κατάρτιση του δικαστικού προσωπικού στα κράτη-μέλη, κυρίω όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο. Παραμένουν ωστόσο αρκετά περίπλοκα ζητήματα. Καταρχάς, η προσφυγή στην διαμεσολάβηση σε σχέση με την επιμέλεια που δεν εξασφαλίζει πάντοτε ε, ε, αμεροληψία. Κίνδυνοι Ορισμένοι δικαστές κρατών μελών να λαμβάνουν αποφάσεις προς όφελος των δικών τους υπηκόους εις βάρος του μέλους οικογένεια που έχει θα γίνει άλλου κράτους είναι βεβαίως ορατή ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκ μέρους της ομάδας ENF δίνω το λόγο στον κύριο Λεμπρετόν. Κυρία Πρόεδρε, η διασυνοριακή απαγωγή παιδιών είναι σοβαρό πρόβλημα. Στη Γαλλία αφορά περισσότερο παιδιά από γάλλο-γερμανικές οικογένειες. Όταν τα ζευγάρια χωρίζουν πολύ συχνά οι Γερμανοί παίρνουν τα παιδιά τους στη Γερμανία ενώ η γαλλική δικαιοσύνη μπορεί να έχει αναγνωρίσει την ε, γονική μέρημνα και επιμέλεια στους Γάλλους γονείς. Πολλούς μήνες βλέπουμε αδράνεια και χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που πια αυτές οι φωνές αγωνίες ακούστηκαν. Η έκθεση ΣΦΙΦΚΑ θα επιτρέψει την ευχερέστερη ανάκτηση των παιδιών από τους γονείς τους, ε, ιδιαίτερα τρία στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Ε, πρώτον, περιορίζονται οι προθεσμίες για την επάνωδο των παιδιών στις 18 εβδομάδες. Δεύτερον, στη ε, κράτη-μέλη προβλέπεται θεσμός ειδικευμένου στην απαγωγή παιδιών δίκαστη. Και τρίτον, κεντρικές αρχές των κρατών μελών θα είναι εγγύηστριες των μηχανισμών αυτών στο κάθε κράτος και γι' αυτό θα υπερψηφίσω την έκθεση ΣΒΙΦΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σταρά Φαραγκούτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως οι αντιδικίες σε διεθνείς ζευγάρια και διεθνείς οικογένειες έχουν αυξηθεί γιατί έχουμε 16 εκατομμύρια διεθνείς οικογένειες 140.000 διαζύγια το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1.800 περιπτώσεις απαγωγής ανηλίκων. Όντως, πρόκειται για ένα θέμα που αγγίζει τον ακρογωνιαίο λίθο ε, του συστήματος, τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Ήταν ε, ευνοϊκός ο κανονισμός γιατί ε, βοήθησε και ενίσχυσε τη δικαστική συνεργασία, αλλά μετά από μερικά χρόνια εφαρμογή του διαπιστώσαμε τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του. Γι' αυτό και ήταν απαραίτητη αναδιατύπωση. Υπήρξαν προβλήματα στη δικαστική συνεργασία, όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους. Προβλήματα με την υποδοχή, με την προστασία του ανηλίκου, την ανάθεση ανηλίκου, η απαραίτητη κατάργηση της διαδικασίας εκτελεστότητας, η εκτέλεση των αποφάσεων. Και επίση η ανασφάλεια του δικαίου που μερικές φορές ε, ε, διαπιστώθηκε και οι μεγάλες καθυστερήσεις που απέβησαν εις βάρος του ανηλίκου γιατί ήδη με το χωρισμό είναι τραυματική η εμπειρία για τον ανήλικο και όταν η διαδικασία είναι χρονοβόρα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν την ασφάλεια δικαίου για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να δώσουμε έμφαση στη διαμεσολάβηση για έναν αρμονικό διακανονισμό και διευθέτηση της διαφθοράς με, της διαφοράς συγγνώμη, με λήψη υπόψη φυσικά του συμφέροντος του παιδιού που είναι αυτό που προέχει εδώ. Και θα πρέπει να είμαστε ε, αποτελεσματικοί και να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού. Ευχαριστώ. κυρία Γκούτελαντ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ. Ένα παιδί δικαιούται να είναι ευτυχισμένο. Δεν θα πρέπει να γίνει ε, θύμα και μάρτυρας ε, της αντιδικίας των γονιών του σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου. Είναι θετικό που ε, Υπάρχουν διεθνείς οικογένειες, αλλά δυστυχώς έχουμε 16 εκατομμύρια διασυνοριακές υποθέσεις γαμικών διαφορών και διαφορών γονικής μέρημνας και 1.800 παιδιά είναι θύματα απαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θύματα σε τελική ανάλυση αυτής της κατάστασης είναι τα ίδια τα παιδιά και γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σχετικό κανονισμό Βρυξέλλες 2α αν θέλουμε το καλό του παιδιού είναι συγκεχημένος ο διαγωνισμός και δημιουργεί μια ανασφάλεια δικαίου. Γι' αυτό και είναι σημαντικό και απαραίτητο να λάβουμε υπόψη το συμφέρον του παιδιού και να μεριμνήσουμε ε, για την προστασία του παιδιού και τη λήψη υπόψη του συμφέροντός του. Ελπίζω να υπερψηφιστεί αύριο η έκθεση. Επίσης θα θέλαμε να καλυφθούν όχι μόνο οι γάμοι αλλά και τα σύμφωνα συμβίωσης και λυπούμε που η συντηρητική απορρίπτω τη συμπερίληψη του συμφώνου συμβίωσης στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Γιατί το υπέρτερο εδώ αγαθό είναι το συμφέρον του παιδιού και αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των προσπαθειών μας. Ο κύριος Μπρανίσλαφ Σκρίπεκ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Σβιέφκα για την έκθεση ε, η οποία αφορά τις ε, περιπτώσεις απαγωγής ε, παιδιών. Οι συνάδελφοί μου συνέβαλαν στο να αναζητηθεί μια λύση. Το διαζύγιο πάντα είναι τραγωδία γιατί επηρεάζει τη ζωή των παιδιών. Οι γονείς ε, που βρίσκονται σε αντιδικία, αυτό δεν είναι σωστό. Ε, θα έπρεπε να είναι γονείς ε, που δείχνουν αγάπη μεταξύ τους. Τα παιδιά πρέπει να εισακούνται, να λένε τη γνώμη τους, σε ποια χώρα θέλουν να ζήσουν, με ποιον γονέα. Όποτε όμως έχουμε και οποτεδήποτε έχουμε απαγωγή παιδιών, διαπιστώνουμε ότι εκεί προκύπτουν τεράστια προβλήματα. Είμαι σίγουρος ότι το κοινοβούλιο αυτό θα λάβει υπόψη του το καλό του παιδιού, θα προστατεύσει τα παιδιά και θέλω να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα και των αγέννητων παιδιών. Κυρία Εύη, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πολλοί είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, που καταγγέλουν ακόμη στην Επιτροπή Αναφορών πολύ σοβαρέ παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους που προσπαθεί ο κανονισμός αυτός και η έκθεσή μας να αντιμετωπίσουν κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό. Πρόκειται για αναφορές οι οποίες κυρίω έχουν να κάνουν με μηχανισμούς, πρακτικές διαδικασίες στην ε, πράξη ε, που εντοπίζονται κυρίως στη Γερμανία σε σχέση με μη Γερμανούς γονείς σε περίπτωση γαμικών διαφορών και επιμέλεια. Οι γερμανικές αρχές ε, ισχυρίζονται ότι είναι διατεθειμένες να δώσουν πλήρη συνεργασία, να συνεργαστούν πλήρως. Βέβαια έχει περάσει πολύ καιρό και ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και έτσι η αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων που μπορούμε να εξασφαλίσουμε χάρη στον κανονισμό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ απλή ε, συνέπεια το ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία και δεν θα χρειάζονται βαριές δικαστικές διαδικασίες, έλεγχοι και επαληθεύσει σε σχέση με τις δικαστικές ή τις άλλες αρμόδιες αρχές στην κάθε χώρα σε σχέση με τις ε, εγγύησεις για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ε, η κυρία Ζάμετ ο κύριος Ζάμετ Τιμέκη. Πρόεδρε, όλοι συμφωνούμε πως ε, πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά από κάθε κίνδυνο και αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ευρωπαϊκών μας αξιών. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν να προσφέρουμε αυτή την προστασία, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο θα διευθετούνται οι περιπτώσεις διεθνών απαγωγών. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σαφέστερα ένδικα μέσα και αυτό το βλέπουμε με μια περίπτωση που ανέκυψε στη Μάλτα. Πατέρας α, Μαλτέζος είχε την επιμέλεια του παιδιού του με αποφάση δικαστηρίου της Μάλτας. Δεν μπόρεσε όμως να επιβάλλει την απάντηση διότι η μητέρα απήγαγε το παιδί και εγκατέλειψε το νησί. Μιλώ για αληθινή περίπτωση, πραγματική περίπτωση που πειράζει βέβαια την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Με τον κανονισμό αυτό λοιπόν θα μπορεί να ε, επιστρέφει στον τόπο κατοικία του το παιδί πολύ σύντομα, σε σύντομο διάστημα, με σύντομες διαδικασίες. Θα προβλέπεται η διαδικασία της διάμεσολάβησης και ταυτόχρονα θα υπάρχουν μέτρα για την επιβολή μιας πολύ απλής αρχής που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, τη διαφύλεξη δηλαδή του συμφερόντος του παιδιού. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, και δίνω το λόγο στην κυρία Κινίτσι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Η πρόταση κανονισμού που συζητούμε ε, έρχεται ως απαραίτητη βελτίωση και επικαιροποίηση του κανονισμού για διάφορα κενά που βλέπουμε συχνά να αναδύονται στα ευρωπαϊκά κράτη σε σχέση με αποφάσεις σε γαμικές διαφορές γενικά αλλά και ιδίως ε, σε περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών όπου είναι πολύ μακροχρόνιες οι διαφωνίες και οι δικαστικές διαφορές μεταξύ των γονέων όταν πρόκειται για διεθνείς περιπτώσεις υποθέσεις. Ε, ιδιαίτερη σημασία έχει η ακρόαση του ανηλίκου για να μπορεί να εκφράσει το ίδιο το παιδί τις επιθυμίες του, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, και να δίνονται στις δικαστικές αρχές όλα τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να αξιολογήσουν ποιο είναι το δικό του υπέρτερο και υπέρτατο συμφέρον. Πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα για την επιμέλεια του παιδιού και κάθε μέτρο και εγγύηση ώστε να μην ανατρέπεται ε, η ηρεμία του, να μην τραυματίζεται το παιδί. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η επιτάχυνση των διαδικασιών για επιστροφή στην αιστεία του του παιδιού, η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων ε, σε ειδικευμένε αρχές μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής και έτσι δεν θα υποβάλλεται σε μακρές περιόδους αβεβαιότητας λόγω της δικαστικής διαδικασίας το παιδί. Συγχαίρω και ευχαριστώ τους συναδέλφους της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων για την εξαιρετική τους δουλειά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ράντεφ. μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Ταντέους Σιβιεύκα, για την αρτιότατη έκθεσή του και χαίρομαι ιδιαίτερος που μεγάλο τμήμα των τροπολογιών μου συμπεριλήφθηκε στην οριστική μορφή του κειμένου και ελπίζω το Συμβούλιο να αφογκραστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λάβει υπόψη τι τροπολογίε του, παρόλο που στην περίπτωση αυτή η διαδικασία που ισχύει για το Κοινοβούλιο είναι απλή διαδικασία διαβούλευση. Ελπίζω παρόλα αυτά ότι με τι προτάσει μα θα συμβάλλουμε στην καλύτερη προστασία του συμφέροντο του παιδιού στα, στην περίπτωση

αρμόδιων φορέων και σε περίπτωση διεθνών ζευγαριών θα πρέπει να ενημερώνονται και οι δύο διάδικοι για τη διαδικασία και τα μέτρα που έχουν, ληφθού, που έχουν ληφθεί εις βάρος τους και μάλιστα στη γλώσσα που οι διάδικοι καταλαβαίνουν καλύτερα. Είναι σημαντικό επίσης να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού και να λάβουμε υπόψη και την εθνοτική, ε, πολιτιστική του και γλωσσική προέλευση. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ανάθεση του παιδιού να αναδίθεται κατά πρώτο ε, στους γονείς του ή στους στενούς συγγενείς, ακόμη και διαμένουν σε άλλη χώρα. Επίσης, θα πρέπει οι γονείς και τα μέλη της οικογένειας του παιδιού να έχουν τακτικές επαφές μαζί με το παιδί του, παρόλο που μπορεί να διαμένουν σε άλλη χώρα. Θεωρώ ότι ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α θα πρέπει να σέβεται τη συναρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα αγωνικής μέρημνας και να μην επιβάλλει στα κράτη-μέλη συγκεκριμένα νομικά μέτρα που δεν συνάδουν με τις παραδόσεις τους. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Πόσπης έχει το λόγο τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα αυτή τη συζήτηση. Ε, κάποια εποχή ήμουν υπουργό δικαιοσύνη στην ε, Τσεχία και ασχολήθηκα με την απαγωγή των παιδιών. Στην πράξη είδαμε ότι δεν λειτουργεί αυτή η συμφωνία και υπήρχαν πάρα πολλά κενά. Ε, χαίρομαι που λύσαμε τα προβλήματα υπήρξε ε, ασαφής θέση πολλών δικαστηρίων. Σε αυτή λοιπόν την εκδοχή ρυθμίζονται όλα τα θέματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή η νέα εκδοχή θα έχει ε, θετικές συνέπειες. Να έχουμε ειδικά δικαστήρια, να υπάρχουν προθεσμίες ε, για δικαστικές αποφάσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν στο να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των παιδιών. Ως κάποιος ο οποίος έχει πρακτική εμπειρία θέλω να πω ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι αυτή η νομική προσαρμογή θα συνεπάγεται πολλά σημαντικά ωφέλη στην πράξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλά, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Πώ θα ήταν δυνατόν να μην έχουμε πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να τάσεται υπέρ, με τέτοια μεγάλη διαφορά, υπέρ ενός κανονισμού που στόχο έχει την ενίσχυση της αρχής της αμοιβαία εμπιστοσύνη και της αμοιβαία αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο θέμα όπω είναι το θέμα γαμικών διαφορών, διαφορών μέρη μα και πάνω απ' όλα απαγωγή παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν αναμενόμενο να έχουμε τέτοια συντριπτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν ήμουν υπουργό ε, δικαιοσύνη στην Ισπανία ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το θέμα αυτό και χαιρετίζομαι αυτή την πρόοδο που στόχο έχει την αποκατάσταση τη ασφάλεια δικαίου, την κατάργηση τη διαδικασία εκτελεστότητας και κυρίω ε, την ενίσχυση των δικαιωμάτων ε, του, των ανηλίκων. Λυπάμαι που δυστυχώ δεν τελεσφόρησαν οι τροπολογίε τη επιτροπή Αναφορών. Εκεί ε, ζητήσαμε την ενίσχυση των δικαιωμάτων του παιδιού σε τόσο τραυματικές και επώδυνες διαδικασίες σε περίπτωση ενδοκογενειακής ή έφυλης βίας ή την έκφραση της οικογένειας, των διαφόρων μορφών οικογένειας που υπάρχουν, συνυπάρχουν και εμπλουτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει χαιρετίζω τον κανονισμό και θα υπερψηφίσω την έκθεση τη Ευχαριστώ κύριο Μαριά, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η αναδιατύπωση του κανονισμού 2201 του δύο για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και σε διαφορές γονικής μέριμνας θεωρώ ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. στην επιτροπή αναφορών είχαν έρθει πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες είχαν σχέση και με την εξάσκηση της γονικής μέριμνας και με απαγωγές μάλιστα είχαμε πάρα πολλέ καταγγελίε για τον τρόπο λειτουργία τη ειδική υπηρεσία πρόνοια στη γερμανία το περίφημο jugendamt και θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβαση του κυρίου γκέρικ και ήθελα να τον συγχαρώ που πραγματικά ζήτησε από την πατρίδα του να υπάρξουν αλλαγέ στο θέμα αυτό. είναι προφανέ ότι ο κανονισμό ε, έχει μεγάλη σημασία διότι επικεντρώνεται στο συμφέρον του παιδιού. θεωρώ σημαντικό ιδιαίτερα τη δυνατότητα Ακρόαση του ίδιου του παιδιού προκειμένου να εκδοθεί συγκεκριμένη δικαστική απόφαση. επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι θεσπίζονται ειδικευμένα δικαστήρια τα οποία εξετάζουν τις περιπτώσεις απαγωγής παιδιών. αυτά είναι τα κεντρικά σημεία και νομίζω ότι βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Συγγνώμη. Πρώτα στον κύριο Μαλάνκα. Μαστάλκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να ακούμε τη φωνή ενό παιδιού όσο μιλάω, ε, μάλλον είναι εδώ παρόν ο γιος της συναδέλφου μου, αν τυχόν ακούσετε τέτοια φωνή. Θέλω λοιπόν να ακούσω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων που έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά για, την, για τα θέματα της επιμέλειας. Ε, είναι πολύ σημαντικό το έργο αυτό, ιδιαίτερα για την περίπτωση των υπερσυνοριακών ε, απαγωγών. Ε, διευκολύνεται η εργασία των αρμόδιων θεσμών και ιδιαίτερα στις απαγωγές από ένα γονιό, γιατί κάθε λεπτό χάνεται στην Ευρώπη ένα παιδί το 2015. Ήταν περισσότερα από 60.000 οι απαγωγές που καταγγέλθηκαν. Με τον ε, καρονισμό λοιπόν σήμερα μπορούμε να βρούμε λύσεις που προστατεύουν το παιδί και καλωσορίζω την προσέγγιση του εισηγητή ο οποίος επέλεξε μια σαφή, ε, έκανε μια σαφή επιλογή. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην κρυπτή. τη ασφάλεια δικαίου που εξασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού και απλοποιεί την έβρεση λύση. Είναι επίση απαραίτητη η διατήρηση του οικογενειακού δικαίου υπό την πλήρη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της υποπροποθέσει δυνατότητα άρνησης αναγνώριση αποφάσεων. Παρ' όλα αυτά, για συναισθηματικά φορτισμένα και πραγματικά ζητήματα επιχειρείται η διατάραξη νομική τάξη και λογική απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της δυτικής νομικής προσέγγισης που αφορά σε λαθρομετανάστες και σε άτομα των οποίων η συνήθις διαμονή δεν μπορεί να διευκρινιστεί οι οποίοι αρνούνται την κοινωνική και πολιτισμική τους εσωμάτωση και έχουν διαφορετικές ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες. σεβόμενοι τις συνθήκες οφείλουμε να περιοριζόμαστε στην υποστήριξη ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών και διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών δίχως εμπλοκή στη διαρρύθμιση της φύσης των οικογενειακών υποθέσεων και με μέλημα το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σαμπόρσκα, έχει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη βελτίωση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την μετώπιση των υπερσυνοριακών γαμικών διαφορών και απαγωγών, με σεβασμό βέβαια των αρμοδιοτήτων ε, των κρατών μελών σε τέτοια θέματα. ώστε να μην παραβιάζεται η ένωμη τάξη των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικές ε, τέσσερις τροπολογίες, δύο εκ των οποίων ζητούν την συνεργασία των κρατών μελών ώστε να αναγνωρίζουν τις ε, ε, ενώσεις προσώπων και επίσης δύο άλλες τροπολογίες έχουν να κάνουν με αποφάσεις δικαστηρίων της Άριας. Χαίρομαι που ο κύριος Σβιέφκα έχει κατά κύριο λόγο στραφεί στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Αλλά σε αυτά δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω. Ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ έχει το λόγο. Τελευταία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στην ιστορική στιγμή που διανύουμε, όταν η κινητικότητα των ατόμων και των μελών της οικογένειάς τους έχει γίνει καθημερινότητα, ε, δημιουργείται μεγαλύτερη ανάγκη για τη θέσπιση νομικών πλαισίων σε όλα τα κράτη, σε επίπεδο κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, έχει νευραλική σημασία να σεβαστούμε τα όρια των κοινοτικών αρμοδιοτήτων και να μην επιτρέψουμε με υπερβολική νομοθετική φιλοδοξία να παραβιαστούν οι αρχέ τη επικουρικότητα και των ε, αποκλειστικών εθνικών αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό και ακριβώς σας ζητώ να καταψηφίσετε τις ε, τροπολογίες 19, 28, 31 και 49. Ε, με την πιθανή υπερψήφιση αυτών των τροπολογιών η δημόσια τάξη των κρατών μελών δεν θα λαμβάνεται πια ε, υπόψη σε περίπτωση ε, γονικής μέρημνας και παραβιάζεται το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουμε το εθνικό του ουσιαστικό δίκαιο τα οικογενειακά ζητήματα. Δεν θα πρέπει να ανατρέψουμε κάτι που αναρρύθμιτες φορές έχει βεβαιώσει ο Ευρωπαίος Δικαστής, δηλαδή ότι η δημόσια τάξη και η δημόσια πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μέλλον. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία Catch the Eye και τώρα μπορούμε... Ή μάλλον ο κύριος Πόλτσακ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Εγώ παρακολούθησα όλη τη συζήτηση και γι' αυτό δικαιούμαι να μιλήσω στο Eye. Αξιότιμη ε, κυρία, αξιότιμη συγητά, ε, Νομίζω ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με μια πραγματική σχηνοβασία, γιατί οι διαδικασίες αυτές υποτίθεται ότι θα βοηθούν στο να αντιμετωπίζονται οι αντιδικίες ε, ανάμεσα στους γονείς. Αυτό που παίζει ρόλο είναι να προστατεύεται το καλό του παιδιού. Αυτό πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας, ε, χωρίς ε, να παρισφρίουν ιδεολογίες. Πρέπει να λαμβάνονται ταχύτατα αποφάσεις, να υπάρχουν και να τηρούνται οι προθεσμίες. Η αναθεώρηση του κανονισμού των Βρυξελών είναι πολύ σημαντική. Εξίσου σημαντικό είναι οι γονείς να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και για τις υποχρεώσεις τους. Και με τον τρόπο αυτό να μπορούν να συμβάλλουν στη διαμεσολάβηση. Όμως αυτός ο κανονισμός δεν αφορά βέβαια τη διαμεσολάβηση. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κύριο Αβραμόπουλο, στον κύριο Επίτροπο. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες μου εκ μέρους της Επιτροπής για την έκθεσή σας και την υποστήριξη για την πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού. Η έκθεσή σας θα εμπνεύσει και τις συζητήσεις στο Συμβούλιο. Είμαστε βέβαιοι ότι υπό τη Βουλγαρική Προεδρία που όρισε ως προτεραιότητα το θέμα αυτό θα δούμε πρόοδο στο θέμα αυτό ταχεία διεκπαιρέωση των ε, συνομιλιών θα, είναι, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα διευκολύνει η οικογένεια σε δύσκολες ε, συνθήκες και θα προστατέψει ιδιαίτερα τα παιδιά. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα οδηγήσει στην υιοθέτηση μέτρων που θα υπηρετήσουν ακριβώς αυτόν τον ευγενή στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και τώρα παρακαλώ τον εισηγητή κύριο Σβιεύκα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους ε, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με την ψηφοφορία αυτή ολοκληρώνουμε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία. Αλλά ελπίζω ότι ο καρπός των εργασιών μας να εγκριθεί και αύριο στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια και να ληφθεί το αποτέλεσμα των εργασιών μας υπόψη και στο Συμβούλιο. Και θα ήθελα να σας ε, καθησυχάσω γιατί από ό,τι ξέρω αύριο δεν θα ψηφίσουμε καμία τροπολογία στην έκθεση γιατί μόνο με μονομένες ε, τροπολογίες θα ψηφίσουμε. Οπότε όσοι μέχρι στιγμής είχαν ε, για να υπερψηφίσουν μπορεί να το κάνουν γιατί όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων με διαβεβαίωσαν ότι θα υπερψηφίσουν ε, την έκθεση. Σε αυτό ε, με διαβεβαίωσαν και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά. Οπότε δεν θα έχουμε τροπολογίες ε, των πολιτικών ομάδων παρά μόνο μεμονωμένες αύριο. Σίγουρα αυτή η διαδικασία στόχο έχει να επιλύσει κάποια προβλήματα της οικογενειακής ζωής. Σε καμία περίπτωση δεν σφετεριζόμαστε, δεν μπαίνουμε στα χωράφια του οικογενειακού δικαίου που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και ούτε η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε η έκθεση δεν παραβίασαν την αρχή της επικουρικότητας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Ε, αυτή η πρόταση θα είναι η λιδία λίθος ε, για την αμοιβαία αναγνώριση και αμοιβαία εμπιστοσύνη των δικαστικών αποφάσεων ε, και των δικαστικών συστημάτων. Χρειάζεται αυτή η εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών συστημάτων και αυτό πραγματικά θα είναι η λιδία λίθος και για την εμπιστοσύνη στα, επόμενα, στα άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ. Και έτσι ολοκληρώνεται.